Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη ε, είναι η έκθεση της κυρίας Ρης για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Το λόγο έχει πρώτα για τέσσερα λεπτά η συγκεκριά μας η κυρία Ρης. Κυρία Ρίς, παρακαλώ, ανάψτε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να χαιρετήσω και την Δανική Προεδρία, αλλά δεν ξέρω την επομένη της ήττας τους απουσιάζουν. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω τους κυρίους Δελόγκ, Ζαρμπούγκου, ε, Γκέρλινγκ, Λεωτάρ, τον Κάρλ Σλέτερ επίσης, ε, που με βοήθησαν ως και όδης συγητές ε, των πολιτικών τους ομάδων και απέδειξαν ότι όλοι από κοινού είμαστε πολύ πιο ισχυροί. Εν τη ενώση ισχύς. Ε, ε, φυσικά συνεργαστήκαμε και για το συμφέρον των οικογενειών, των ευάλωτων, των ευπαθών ανθρώπων και κυρίως όσων ενδιαφέρονται από την νομοθεσία αυτή που αφορά ειδικά τρόφιμα. Το κείμενο αυτό είναι σημαντικό για τα βρέφη, τα παιδιά κάτω των τριών ετών και τους μακροχρόνια άρρωστους που χρειάζονται ειδικές τροφές, έχουν ειδικές διαιτητικές ε, ανάγκες. Έχουμε τρόφιμα συγκεκριμένου κοινού που καλύπτουν 2%, ένα ιδιαίτερα επαθές κοινό, 2% της τεράστιας ε, αγοράς των τροφίμων ξεκινήσω με τις απαρχές αυτής της νομοθετικής πρόταση. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευτυχώ μετά από 35 χρόνια εφαρμογή νομοθεσία για τις διαιτητικέ τροφές και οι διάλε ειδικέ τροφές πρότεινε πλήρη μεταρρύθμιση αυτής της ε, ιδιάζουσας νομοθετικής ε, ε, διάταξης. Θα πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτά τα τρόφιμα γιατί ε, αυτή η αταξία δημιουργεί προβλήματα στην εσωτερική αγορά και πολύ συχνά δεν επιτρέπει στον καταναλωτή να ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερη επιλογή. Με την ομόφωνη ψηφοφορία που είχαμε στι 29 Φεβρουαρίου για την έκθεσή μου, η Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, ε, έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα και σαφέστατο μήνυμα. Και μάλιστα η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση της νομοθεσία αυτής και για την κατάργηση της έννοια τη διαιτητική στροφή είναι πολύ σωστή και την υποστηρίξαμε. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο ε, συγκεκριμένα για τρία, για τρία είδη τροφών, για, τα, για τις τροφές και των μικρών παιδιών και τις τροφές για αρρώστους. Πρόκειται για υπομάδες, ευπαθείς υπομάδες πληθυσμού που δεν μπορούν να ασκήσουν την ελεύθερη επιλογή τους. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό για μας να θεσπίσουμε αυστηρούς κανόνες και για τη σήμανση και για τη σύνθεση αυτών των τροφών. Επίσης, θελήσαμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής προκειμένου να περιλάβει και άλλε ομάδες, ε, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Για παράδειγμα, όσους έχουν ε, υπέρβαρο, όσους έχουν, από ε, παχυσαρκία και πρέπει να καταναλώνουν ε, χαμηλές τρόφιμα με χαμηλές θερμίδες και όσους πάσχουν από κοιλιοκάκι και δυσανεξία γλουτένης. 2% του κοινοτικού πληθυσμού υποφέρει από αυτή την ασθένεια και είναι υπέρ του ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη. Θα ήθελα να σα επιθυμίσω ότι η νομοθεσία αυτή στόχο έχει να προστατεύσει του πιο ευπαθείς από εμά, τους πιο ευάλωτους. Είναι κέρια σημασία. Επίσης δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα εδώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και τις πιο δυναμικές μας επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσει που αποτελούν την καρδιά τη καινοτομία και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ε, ιταλικές αυτές, βελγικές, ε, γερμανικές εταιρείες. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φυσικά ήρθαν σε επαφή μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης έκθεσης με αρκετές ανησυχίες γιατί με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούνται κάποιες αλλαγές στον κανονισμό του 2006 για τους ισχυρισμούς. Νομίζω ότι το σημαντικό επιχείρημα είναι το κόστος που θα πρέπει να αναλάβουν για να υποβάλουν στην ΕΦΣΑ εντοσχέ κόστους 500.000 ενός ευρώ για να τεκμηριώσουν τα αιτήματά τους για συγκεκριμένες τροφές. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσουμε ε, θεμητό ανταγωνισμό. Η πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι εγκάρσια σε όλη μας την νομοθεσία. Θα πρέπει να το επιθυμίσουμε εδώ. Ένα σύντομο μήνυμα προς τους και οδησηγητές. Θα Καταλάβατε ότι εγώ ως συγγήτρια θα πρέπει να εμείνω στις συνολικές συμβιβαστικέ λύσεις, ε, όπως προέκυψαν από την Επιτροπή. Δεν θέλω να ανοίξω νέα μέτωπα και να ξανανοίξουμε συζητήσεις. Μπορεί προσωπικά να είμαι υπέρ κάποιων τροπολογιών, της 84 για παράδειγμα, για τα φυτοφάρμακα, αλλά παρόλα αυτά θα εμείνω στην ε, συνολική συμβιβαστική συμφωνία μας, που καλύπτεται από την ε, τροπολογία 63. Άλλωστε, ο λόγος πρέπει να τηρείται και δεν θα πρέπει να θετείτε. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρης. Εκ μέρους της αρμόδιας καθήλη επιτροπής και για τρία λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Ντάλι. Όχι, όχι, ε, διορθώνει ο πρόεδρος. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει ο Επίτροπος Ντάλι. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σε ευθυγράμμιση με την αρχή για καλύτερη ε, ε, διευθέτηση νομοθετικά των θεμάτων, ε, ο κανονισμός για, την, για τα πρόθυμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά προσπαθεί να ξεπεράσει κάποια αμφιλεγόμενα σημεία. Λαμβάνουμε υπόψη μας αυτούς τους, τους ειδικούς πληθυσμούς και αυτός είναι ο κύριος στόχος της πρότασης που συζητούμε σήμερα. Πριν ασχοληθώ με την ουσία της πρότασης, ε, θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Ρίσε, η οποία προετοίμασε την έκθεση αυτή και βεβαίως και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφέρω ότι και η ΙΜΚΟ και η ΙΤΡΕ συνέβαλαν ε, στην εκπόνηση της εκθέσεως αυτής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται με το εύρος των προτινόμενων τροπολογιών. Η ιδέα της κατάργησης των διαιτητικών ε, ε, τροφίμων ε, είναι μια καλή ιδέα και θα δώσει τέλος σε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας το εύρος ε, της, του προτινόμενης νομοθεσίας ε, θα αφορά συγκεκριμένες ε, κατηγορίες τροφίμων που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού. Συγκεκριμένα βρέθηκε και μικρά παιδιά, καθώς επίσης και ανθρώπους που χρειάζονται ειδική διατροφή για ειδικού ιατρικούς σκοπούς. Κάποιες από τις προτινόμενες τροπολογίες προτείνουν να προσθεθούν κάποιες διαιτητικές ε, τροφές ε, παρότι πιστεύω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους οριζόντιους κανόνες των τροφίμων ε, κατανοώ τον προβληματισμό του Κοινοβουλίου και μπορώ να δεχτώ την συμπερίληψη εδώ όμως δεν μπορώ να δεχτώ τα προϊόντα χωρίς γλουτένι Πιστεύουμε ότι η συμπερίληψη αυτή αφενός δεν είναι απαραίτητη, ε, αφετέρου ε, δεν ε, μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς που πάσουν από κοιλιοκάκι. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι κανόνες που ήδη υφίστανται για αυτά τα τρόφιμα. Αλλά θα πρέπει με καλύτερο και απλούστερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό ε, βάζοντας όλα τα στοιχεία αυτά στον κανονισμό για την ε, πληροφόρηση όσον αφορά τα τρόφιμα. Ε, και επίσης για τα προϊόντα που δεν είναι ήδη προσκευασμένα θα πρέπει να μπουν και αυτά στην ίδια κατηγορία έτσι ώστε η προστασία να είναι γενικότερη. Ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, οι οποίες αφορούν τη μειωμένη χρήση εντομοκτώνων ε, για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ συμμερίζομαι το προβληματικό και την ανησυχία του Κοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των βρεφών και των μικρών παιδιών και όλες οι προσπάθειές μας προς τα εκεί Πρέπει να σας πω όμως ότι οι λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα πρέπει να δοθούν σε εξουσιοδότηση πράξη. Ε, την ίδια θετική προσέγγιση έχω και όσον αφορά την προετοιμαστία ε, έκθεσης ε, για τροφές για αθλητές και για ηθικά γάλατα για νεογνάμ. Πιστεύουμε ότι μέσω ε, πράξεων κάτε ε, εξουσιοδότηση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, και όχι με εφαρμοστικές πράξεις. Υπάρχουν κατά αυτή την έννοια οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Όσον αφορά την Without Όσον αφορά τη διαφήμιση, πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση είναι δυσανάλογα αντίστοιχη ε, με το πεδίο της ε, πρότασης ε, και επομένως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην καλή λειτουργία της αγοράς. Όπως βλέπετε είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία μας ενώνουν περισσότερα από ό,τι μας χωρίζουν και είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα οδηγήσει σε μια ε, ε, έφορη δεύτερη ανάγνωση. Ε, αυτά και θα είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας τώρα και για ένα λεπτό το λόγο κύριο Στάκουλα. Kiitoksia arvoisa Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα ε, να ευχαριστήσω την κυρία Ρή στην για την εξαιρετική εργασία. Ε, έκανα την ε, ε, το γνωμοδότηση, συνέταξε τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ίντα και ήταν πολύ εύκολο έργο διότι χρειαζόντουσαν νέες διατάξεις καθότι η παλαιά νομοθεσία ήταν όντως πεπαλαιωμένη και πρόκειται για τρόφιμα για παιδιά και για ειδικού στόχους όπου πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση πάνω στην συσκευασία το κείμενο πρέπει να είναι κατανοητό, σαφές ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διατυπώσεις οι οποίες μπορεί να παραπλανήσουν πρέπει ο πολίτης και καταναλωτής να γνωρίζει τι καταναλώνει. Θέλω να σας πω ότι γνωρίζω και προσωπικά τον τομέα των τροφίμων. Χρησιμοποίησα και εγώ αυτά τα τρόφιμα όταν μεγάλωνα και δεν πρέπει να υπάρξουν παρανοήσεις. Ευχαριστώ κύριε Ταχούλα. Εκ μέρου τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και για ένα λεπτό, το λόγο έχει η κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν πολλά προσόντα από αυτή την νομοθεσία που θα προστατεύσει πιο αποτελεσματικά τους καταναλωτές. Η σήμανση πρέπει να είναι σαφής και δεν πρέπει να παραπλανεί. Ε, Παραδείγματο χάρη πρέπει να ξέρουμε πότε δεν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση ένα τρόφιμο διότι μέχρι στιγμής δεν είναι τελείως σαφές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει προστασία για τις ευάλωτες ομάδες δηλαδή ε, τα ε, γάλατα για βρέφη και παιδιά ε, πρέπει να παρουσιάζουν όλη τη σύνθεσή τους και να γνωρίζουμε εάν βοηθούν στην ανάπτυξη των παιδιών. Πέραν αυτού όμως θα χρειαστεί μια καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που θα επιτραπεί μέσω αυτής της νομοθεσίας για να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και ελπίζω ότι θα υπάρξει και μία ισορροπία για να βοηθηθεί η υγεία των καταναλωτών και ευχαριστώ για τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Ευχαριστούμε κύριε Ιβάνομα. Ιβάνοβα. Περνάμε στους ομιλητές ε, των ομάδων. Για 1,5 λεπτό από το ΕΛΚ, κυρία Ντελάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρους του ΕΛΚ να συμφωνήσω με την εισηγητρία και να ευθυγραμμιστώ με τη θέση της, επενώντας την για το έργο της. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί η σχετική νομοθεσία, γιατί υπάρχουν πολλά τρόφιμα ειδικού προορισμού και θα πρέπει η νομοθεσία να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, προσπαθώντας να προστατεύσουμε ταυτόχρονα τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε ειδικό καθεστώς για τις ειδικέ ε, τροφές που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς, για τις βρεφικές τροφές των παιδιών, καθώς και τις διαιτητικές τροφές, ιδιαίτερα τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη για τα άτομα που πάσχουν από δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπαχθούν αυτά τα τρόφιμα στη Γενική Νομοθεσία. Εμείς ε, ε, κάναμε το καθήκον μας. Ε, με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίναμε την έκθεση της κυρίας Ρης. Φαντάζομαι ότι θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία και στην Ολομέλεια. Το μπαλάκι είναι τώρα στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη διαπραγματευτική εντολή και να καταλήξει σε μια συμφωνία. Γιατί έχουμε το, γάλα, το γάλα πρώτης βρεφικής και δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Τι θα γίνει, με, πώς θα χαρακτηριστεί αυτό το προϊόν που είναι θεμελιώδες για ένα μικρό παιδί και φυσικά είναι θεμελιώδες το βρεφικό γάλα και για τα βρέφη. Τι γίνεται με την περιεκτικότητα σε βιταμίνες, με τον εμπλουτισμό. Ποιο γάλα είναι κατάλληλο και ποιο ακατάλληλο. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς νομοθετικές διατάξεις για να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι διαβήτη για παιδιά που θα καταναλώσουν σε πολύ μικρή ηλικία κατάλληλο Αλλά παρακαλώ να διαθετηθούν αυτά τα θέματα το συντομότερο δυνατό. Θα σας είναι ευγνώμονε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει η κυρία Σάρμπου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι έλαβε υπόψη της όλες τις συστάσεις ε, τις οποίες τις υπέβαλαν ε, οι συνάδελφοί της ε, και στην εκπόνηση της έκθεσης και στην ανάλυση των τροπολογιών. Κατά την άποψή μου, Σκοπός ε, αυτής ε, της οδηγίας ε, είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη σωστή πληροφόρηση έτσι ώστε να καταναλώσουν τελικά τη σωστή τροφή. Τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε η νομοθεσία και είναι γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη προστασία του καταναλωτή. Ε, όμως η νομοθεσία για τα διαιτητικά τρόφιμα αποτελούσε πρόσκομα και γι' αυτό Χαιρόμαστε για την πρόταση της Επιτροπής και τις βελτιώσεις που πρότεινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, ένα από τα προβλήματα που είχα ήταν η διαφήμιση ε, και οι ε, σημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά. Πέρα από οποιοδήποτε κανονισμό, τα προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο επιθετικής διαφήμισης υπάρχουν ακόμα μητέρες ε, οι οποίες προσπαθούν να θυλάζουν τα παιδιά τους αλλά το ποσοστό ε, είναι μικρό. Πρέπει να ε, δώσουμε την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν σωστή τροφή και να σταματήσει η δυνατότητα των εταιριών να περιγράφουν αυτές τις διατάξεις. Δεν υπάρχει πάντως καμία ε, ε, καμία απόδειξη ε, ότι τα προϊόντα τα οποία διαφημίζονται ως διατηρητικά προϊόντα είναι καλύτερα από άλλα ή ότι το γάλα το οποίο διαφημίζεται σαν ειδική διατροφή είναι καλύτερο από άλλα γιατί άλλωστε δεν καλύπτει ειδικού ιατρικούς σκοπούς και επίσης οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν τη σήμανση ειδικά για αθλητές ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγήσουν την ε, σήμανση αυτή. Έχουμε δικαίωμα για καλύτερη ε, τροφή. Έχετε μια μπλε κάρτα, τον κύριο Ρούμπιχ, τη δέχεστε. Ναι, βεβαίως. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Σάμπου. Σε αυτή την νομοθεσία υπάρχει και πάλι μεγάλη γραφειοκρατία η οποία συνδυάζεται για τα φυτοφάρμακα. θα ήθελα να ξέρω λοιπόν εφόσον θέλουμε να αποφύγουμε επικάλυψη της νομοθεσίας στην Ευρώπη ε, και υπάρχει ήδη ισχύουσα νομοθεσία γιατί εδώ θα πρέπει να ε, ε, να επαναλάβουμε διαδικασίες που ήδη είναι ρυθμισμένες. Η κυρία Σέρβο, ακριβώς διότι η ισχύουσα νομοθεσία έχει ορισμένα κενά τα οποία εκμεταλλεύονται ορισμένη ορισμένη παραγωγή Χρειαζόμαστε λοιπόν νομοθεσία η οποία να είναι πιο αυστηρή και η οποία θα μπορέσει να εφαρμοστεί κατά τρόπον όλα να είναι σαφέστατα και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη λύση που όλοι επιζητούμε. Ευχαριστώ. Εκ των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, για δύο λεπτά, το λόγο η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της και για τις καλές συμβιβαστικέ προτάσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με τα τρόφιμα ε, είναι ε, και ε, τα τρόφιμα για άτομα με ειδικέ ιατρικές ανάγκες αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Βεβαίω το υποκατάστατο γάλακτος πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδική νομοθεσία σχετικά με τη σύσταση αυτών των τροφίμων για να προστατευτούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Το γάλα για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχει απασχολήσει επανειλημμένως στην ε, Επιτροπή μας και τώρα υπάρχει μία ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα αυτή της νομοθεσίας αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση αυτών των προϊόντων και να προβεί στην διατύπωση ειδική ε, νομοθεσία για τα βρέφη μεταξύ 12 και 16 μηνών κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι κανόνες και ακρίβεια ε, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση που έγινε επί του ε, τους, διότι το συμφέρον των παιδιών προέχει. Κυρία Παρβάνοβα, υπάρχει μία μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Σλίτερ. Την δέχεστε. Κύριε Σλίτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώς ήθελα να σας πω ότι εγώ ο, μιλώ ο, εν ονόματι της ομάδος των Πρασίνων και όχι η κυρία Ριβαζή. Αυτό απλώς ήθελα να σας πω. Εντάξει. Ε, κυρία Παρβάνοβα μπορείτε να ηρεμήσετε. Ο κύριος Σλίτερ δεν έχει εχθρικές προθέσεις εναντίον σας. Έχετε το λόγο τότε κύριε Σλίτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την κυρία Παρβάνοβα συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Αλλά θα μιλήσω σου ειδικά. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους ευάλωτους καταναλωτές πράγμα το οποίο ε, επιτυγχάνουμε μερικώς με την απλοποίηση των κανόνων αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ε, οι περιορισμοί στην διαφήμιση για το βρεφικό γάλα υποκατάστατο του θυλασμού και νομίζω ότι χρειάζονται να έχουμε ε, πλέον σοβαρούς ε, κανόνες για τα εντομοκτώνα. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε εντομοκτώνα στην παραγωγή τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ε, την διατροφή των βρεφών. Θα πρέπει επιπλέον να έχουμε ειδικέ κατηγορίες φαρμάκων και γι' αυτό ελπίζω ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να βρουν μία ικανοποιητική λύση για όσους είναι δυσανεκτικοί εις ε, την ε, γλουτένη αλλά και στη σόγια και σε άλλες ουσίες και ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές για δύο λεπτά το λόγο κυρία Γκέρλινγκ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια, καθώς επίσης και στους σκιώδες. Η καλύτερη νομοθεσία πρέπει να απλουστεύει και την ίδια την νομοθεσία και την εφαρμογή τη. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και μέσω και της πρότασης ε, της Κομισιόν. Συμφωνώ ότι ε, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και ε, άνθρωποι με ειδικέ συνθήκε θα πρέπει να έχουν καλή πληροφόρηση. Αλλά αναρωτιέμαι καμιά φορά μήπως μπερδεύουμε περισσότερο την νομοθεσία σε άλλες περιπτώσει αντί να την απλωστεύουμε. Ναι, η συγγήτρια είπε ότι υπήρχε ε, κάποια συμφωνία. Υπήρχε συμφωνία η οποία όμως διεράγει ε, από τη στιγμή που επέμεινε να φτάσουν κάποιες τροπολογίες στην Ολομέλεια. Πρέπει να πω ότι τελικά εγώ δεν προσυπέγραψα την, ε, τον συμβιβασμό πρώτον για τα τρόφιμα που δεν έχουν γλουτένι. νομίζω ότι θα πρέπει η Κομισιόν να βοηθήσει την, τα, τα άτομα αυτά και Βεβαίω εδώ δεν πρόκειται για προστασία των καταναλωτών, πρόκειται για προστασία κάποιων παραγωγών και κάποιων εθνικών διαδικασιών. Αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Επίσης έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με ε, την διατροφή με χαμηλέ θερμίδε και πολύ χαμηλέ ε, θερμίδε. Δεν υπάρχει καμία ε, επιστημονική απόδειξη ότι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικά ιατρικά προβλήματα θα βοηθηθούν αν ε, γίνει πιο δύσκολη η πρόσβασή τους σε προϊόντα τα οποία θεωρούν ε, καλά για την υγεία τους και τους βοηθούν στην κατάστασή τους. Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα του γάλακτος. Βεβαίως ε, υπήρξε μια συγκινησιακή αντίδραση, αλλά δεν υπάρχει καμία ε, επιστημονική απόδειξη ότι με τον τρόπο που ενεργούμε βελτιώνουμε την ε, κατάσταση. Ήδη, κατά την άποψή μου, υπάρχουν ήδη καλοί κανόνες όσον αφορά την χρήση φυτοφαρμάκων. Πέρα από προσωπικές γνώμες, δεν δεν ε, έχει ε, ε, παρουσιαστεί καμία, κανένα ειδικό αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά το θέμα αυτό. Και εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε παρά να προσπαθούν διαρκώς να μας πείσουν, να μας δώσουν τα σωστά επιστημονικά στοιχεία. Κυρία μου, υπάρχει μία μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Γκέρμπερ. Τη δέχεστε? Ωραία. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Γκέρλινγκ διότι μόλις είπε ότι οι ρυθμίσεις για τη δυσανεξία της γλουτένης δεν βοηθούν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα άτομα που πάσχουν από αυτή την πάθηση διότι εάν δεν περιληφθεί ε, εδώ αυτή η διάταξη και υπάρχει μόνο στην διατροφική αλυσίδα δεν θα πετύχουμε το στόχο μας και εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο όπως πρεσβεύει η ομιλήτρια. Η απλή, ε, ε, η απλή απάντηση είναι ότι ε, όντως έχετε δίκιο. Αυτ... Μόνο? Τίποτα άλλο? Το θέμα είναι αν θα βοηθήσουμε ή όχι αυτές τις ομάδες. Εγώ δεν πιστεύω ότι βοηθάμε αυτές τις ευπαθείς ομάδες με την επιπλέον πρόταση. Δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου αυτή η πρόταση. Και ο κανονισμός που προσπαθούμε να καταρτήσουμε ε, για τους χειρισμούς υγείας, ε, τις, ε, τους διαφημίσεις, ο ισχύων κανονισμός ήδη αρκεί. Η συγκεκριμένη πρόταση όχι μόνο δεν θα βοηθήσει, αλλά μπορεί να επιτείνει τη σύγχυση κατά τη γνώμη μου. Καλώ. Εκ μέρου τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κ. Τσιμάνσκι. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μα ε, για τι προσπάθειε που κατέλαβα. Σε ό,τι αφορά το νέο κανονισμό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μέχρι τώρα διατάξεις ε, ε, δεν εφαρμόστηκαν εμπράκτο και έτσι δημιουργήθηκε εύκολη διακίνηση αυτών των προϊόντων με μία εναρμονισμένη και ασαφή νομοθεσία που δημιούργησε στρέβλωση του εμπορίου στο, στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τις αλλαγές που αέρουν τα υπερβολικά διοικητικά εμπόδια και διευκολύνουν την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κυριαρχούν σε, αυτή την ειδικευμένη, σε αυτόν τον ειδικευμένο κλάδο της επισητιστικής βιομηχανίας. Βέβαια το πιο σημαντικό θέμα εδώ είναι το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, ιδιαίτερα όταν οι τροφές αυτές αφορούν πολύ ευπαθείς πληθυσμούς, όπως είναι τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την ε, γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής ε, Επιτροπής που ζητά να, να διευκολυθούν τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν ε, εθνικές διατάξεις στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δικαιολογείται από λόγους προστασίας δημόσιας υγείας. έτσι. Βέβαια δεν θα έχουμε παρόμοια αντιμετώπιση όλων των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσιμάνσκι. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ και Σκανδιναβικής Αριστεράς για 1,5 λεπτό το λόγο η κυρία Σόουζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα όταν μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ και ρίχνουμε μια ματιά στα ράφια με τα γιαούρτια είναι σαν να μπαίνουμε σε φαρμακείο. τόσε υποσχέσει βλέπουμε. Είναι υπερβολική αυτή η διαφήμιση και έρχεται σε αντίθεση βέβαια με την έλλειψη σωστής ενημέρωσης που έχουν ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμοί με ειδικές ανάγκες ε, όσοι έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, τη λακτόζη, διαβητική. Πολύ πιο σοβαρή επίσης είναι η διάθεση αυτών των τροφίμων. Δεν υπάρχουν αυτά τα τρόφιμα εύκολα προσιτά. Μπορεί κανείς να γυρίζει σούπερ μάρκετ και μαγαζί και να μην βρίσκει τα τρόφιμα που χρειάζεται. Ε, οπότε δεν είναι επιλογή αυτή για κάποιον που στερείται οποιοδήποτε επιλογή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η τιμή. Κατά κανόνα αυτέ οι τροφέ είναι πολύ πιο ακριβέ από τα υπόλοιπα τρόφιμα και για ανθρώπους που έχουν ειδικέ διατροφικές ανάγκες, που δεν υπάρχει επιλογή, αλλά ανάγκη θα πρέπει να διευκολυνθεί η αγορά τους με χαμηλότερες τιμές. Δεν θα, μπορούμε, θα πρέπει να δημιουργούμε και εδώ χάσμα μεταξύ αυτών που δίνανται και αυτοί, αυτών που δεν δίνανται να αγοράσουν τρόφιμα που είναι απαραίτητα για τη ζωή τους. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των δικών μας ανησυχιών. Είναι θέμα και δημόσιας υγείας. Και φυσικά οι δράσεις ε, δεν θα πρέπει να επαφεθούν στις λίγες και ισχυρότερε πολυεθνικές της επιστημιστικής βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες που θα πρέπει να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν επιλογή. Είναι σημαντικό για μας η Ευρώπη να μην θυσιάσει την υγεία των πιο ευπαθών ομάδων της. Ευχαριστούμε κυρία Σόουζα. Περάμε στους λοιπούς ομιλητές. Για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ τη Φρεντερή Κρίς για την ε, εκπόνηση της ε, εκθέσεως, αλλά ευχαριστώ επίσης και τη σκιώδη συγγήτρια Έστερ Ντελάντε που εκπροσώπησε πολύ σωστά την πολιτική μας ομάδα. Νομίζω ότι επετεύχθη μια καλή συνένεση στην Επιτροπή και ιδίω ε, σχετικά με την τροπολογία που αναφέρεται εις τους ε, αρρώστους ε, είναι πολύ ε, σωστή η διατύπωση και δεν πρέπει μόνο τα τρόφιμα να μην περιέχουν γλουτένι αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία ισοσκελισμένη σχέση διότι δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς για να μην φάει γλουτένι να μην τρέφεται υγιεινά. Επίσης όσον αφορά τα τα βρέφη και τα ε, παιδιά νεαράς ηλικία ε, θα πρέπει να μην δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε τώρα τη διαφορετική άποψη σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων ή ε, την διατροφή των βρεφών διότι ήδη τη δεκαετία του 90 είχαμε θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα και είχαμε προβλέψει ότι στα βερφικά τρόφιμα πρέπει κανείς να επιτύχει μόνο ότι, να, περιλάβει κανείς μόνο ότι ε, είναι κάτω από το όριο που είχαμε θέσει. Έχω δουλέψει σε ε, νοσοκομείο παιδιατρικό και έχω δει τι ε, πρεσβεύουν οι ειδικοί, οι παιδίατροι, οι οποίοι λένε τώρα ότι αυτά τα οποία προτείνει η κυρία Ρης και άλλοι στην Επιτροπή και άλλοι είναι ρεαλιστικά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής επ' αυτού, ε, διότι ε, για τα ειδικά τρόφιμα πρέπει να υπάρχει ισορροπία και δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι ορισμένοι προστατεύουν καλύτερα τα παιδιά από ό,τι άλλοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότε τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους και όδης εισηγητές και την εισηγήτρια διότι η έκθεση αυτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, υπερψηφίστηκε με 68 ψήφους δηλαδή ε, χωρίς 62 ψήφους δηλαδή ε, σχεδόν ομόφωνα και αυτό δίνει το σήμα ότι θέλουμε υψηλή υψηλό επίπεδο προστασίας ε, και ε, για τον καταναλωτή και για τις εμπλεκόμενες κατηγορίες ε, και ιδίως για τα παιδιά, για τα βρέφη, για τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει πρόβλημα. Έχω δύο παιδιά σε παιδικούς σταθμούς που έχουν αλλεργίες και πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν προσεκτικά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο Ρώση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, να ε, διαγράψει την ιδέα των διατηρητικών προϊόντων ε, ζημιώνει τις κατηγορίες των ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν αυτές τις τροφές, δηλαδή βρέφη, παιδιά μικρής ηλικίας, αθλητές κλπ. Ε, στην Επιτροπή ΕΜΒΗ ε, η άποψη ήταν διαφορετική και επετεύχθη συμφωνία ε, στη, σε πρώτη ανάγνωση και υπάρχουν κάποιες εξαιρέξεις όσον αφορά τα μωρά τα οποία έχουν γεννηθεί προώρα, αυτούς που έχουν τις ανεξίες σε γλουτένη, καθώς επίσης και κάποιες άλλες ειδικέ κατηγορίες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευθετηθούν καλύτερα οι τροφές για για τους αθλητές. Επίσης, για αυτούς που πάσχουν από κοιλιοκάκι θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη. Επίσης, σε μια απλή αναφορά σε λογιογόνους παράγοντες δεν ε, μπορεί να διασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ για 1,5 λεπτό η κυρία Γκροστέτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να απλουστεύσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό είναι πολύ καλό, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει προς ζημία της διατροφικής ασφάλειας και επίσης ε, δεν θα πρέπει ε, να ε, μας απομακρύνει από την διπλή ασφάλεια, δηλαδή υγειονομική και διατροφική κυρίως τον αφορά ευαίσθητες ομάδες, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μιλάμε τώρα για βρέφη, για μικρά παιδιά, για διαβητικούς, για ανθρώπους που θέλουν ειδική διατροφή χαμηλών θερμίδων, ανθρώπους με δυσανεξία στη γλουτένη κλπ. Ε, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις ανεξία στην Λουτέινη ή αυτοί που ακολουθούν ε, ε, διατροφή με χαμηλές θερμίδες δεν κατανοούν την έννοια αυτών που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλουμε ε, να επανισάγουμε τα προϊόντα χωρίς ε, γλουτένη έτσι ώστε να προστατευτούν καλύτερα οι καταναλωτές. Γιατί διαφορετικά η εξαίρεση και η εξαίρεση και η εισαγωγή βαριών διαφορετικών κανόνων δεν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επίσης τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το γάλα συγκεκριμένα για παιδιά από ε, ενό έτου έω ε, τριών, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα πρέπει να ε, αποτελούν μια ειδική κατηγορία, γιατί τα παιδιά αυτά να μην πρέπει να έχουν το καλύτερο γάλα. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό, κυρία uh, Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή ήταν ένα τιτάνιο έργο και χαίρομαι για τι αλλαγέ που πρότειναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Συγγετρία. Θα επικεντρωθώ σε ένα ειδικό ζήτημα που αφορά τη διαφήμιση της, ε, για, τα, για το υποκατάστατο μητρικό γάλα μέχρι 6, για παιδιά μέχρι 6 μηνών. Ε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πιστεύει ότι αυτές οι φόρμουλες δεν είναι ε, Απαραίτητε. και υπάρχει και απαγόρευση για διαφήμιση τέτοιου υποκατάστατο μετρικού γάλακτος. Βέβαια, το γάλα δεύτερη ε, ε, βρεφικής ηλικία επιτρέπεται να διαφημίζεται. Εγώ προσπάθησα να προτείνω επέκταση απαγόρευση, απαγόρευσης, αλλά δεν συγκεντρώσαμε την απόλυτη πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να μπλοκάρουμε αυτόν τον ισχυρισμό τη υγεία. Ε, εξαιτία τη διαφήμιση ε, πολλοί γονεί γνωρίζουν ε, τι διαφορέ μεταξύ του γάλακτο πρώτη βρεφική και δεύτερη βρεφική ηλικία. Ξεκινούν να γάλακτος γάλακτο δεύτερη βρεφική ηλικία υπερβολικά νωρί. Δημιουργείται ένα κενό επειδή το πρώτο πρώτης βρεφικής ηλικίας γάλα επιτρέπεται και το δεύτερης βρεφική ηλικία γάλα απαγορεύεται συγγνώμη, να διαφημιστεί, ενώ το δεύτερη βρεφική ηλικία επιτρέπεται να διαφημιστεί. Έτσι μπερδεύονται οι γονεί και δεν έχουν τεκμηριωμένε αντικειμενικέ πληροφορίε από εμπειρογνώμονε. Δεν θα πρέπει να γίνονται θύματα των βιομηχανιών και να αγοράζουν οι γονεί γάλακτα που δεν είναι απαραίτητα ή δεν είναι κατάλληλα για τα παιδιά του. Θα ήθελα να παροτρύνω του ευρωβουλευτέ να υπερψηφίσουν την τροπολογία 86. Κυρία Γουίλμοντ, η κυρία Ντελάνγκε θέλει να σα υποβάλει ερώτηση με μπλε κάρτα. Συμφωνείτε? Κύριε Ντελάνγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο και πόσος καιρός πέρασε από τότε που χρησιμοποίησε το Formula Milk η κυρία Wilmot αλλά εκεί αναφέρεται το 0 μέχρι 6 μήνε για το πρώτο τη βρεφική ηλικία γάλα. Στο δεύτερο δεύτερης ηλικία ηλικίας είναι από 6 με 12 μήνες. Υπάρχουν μεγάλα γράμματα. Πόσο ε, χαζή πιστεύει η κυρία Γούλμα ότι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε και δεν μπορούν να διαβάσουν 0 έω 6 ή 6 έω 12. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια και να επικεντρώνεται σε, σε λάθος πράγματα. Πιστεύω ότι η τροπολογία 86 είναι περίτη και παρακαλώ να την καταψηφίσετε. Κυρία Γουίλμοντ. Έχετε δίκιο ότι πάει πολύ καιρό που είχα παιδί και είμαι πολύ πιο μεγάλη σε ηλικία από την κυρία που ρώτησε. Και μάλιστα εγώ δεν, χρησιμοποίησα καν ε, γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας ε, γιατί εγώ θύλασα. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Το θέμα δεν είναι αν θα διαλέξει μια γυναίκα να θυλάσει το παιδί της να αγοράσει υποκατάστατο μητρικό γάλα. Αυτό είναι δική της επιλογή. Και Απόλυτο θεμητή, γιατί ο καθένα έχει διαφορετικέ εμπειρίε, διαφορετικού τρόπου ζωή και διαλέγει ό,τι θέλει. Άλλωστε, μπορεί μερικέ γυναίκε να έχουν πρόβλημα με το θυλασμό. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί γονεί, και το απέδειξαν και έρευνε, ότι πολλοί γονεί μερικέ φορέ δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ του γάλακτο πρώτη βρεφική ηλικία και γάλακτο δεύτερη βρεφική ηλικία. Δείτε τι έρευνε αν δεν με πιστεύετε. Δεν θα πρέπει να συμβάλλουμε στην παραπλάνηση των γονέων ε, προκειμένου να αγοράσουν προϊόντα που δεν είναι απαραίτητα ή δεν είναι και κατάλληλα μερικές φορές για τα παιδιά τους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού είναι πολύ σημαντικό χρέος μιας κοινωνίας. Γι' αυτό και ο κανονισμός αυτός για τις τροφές ε, για βρέφη και μικρά, παιδική, και μικρά παιδιά ή για ανθρώπους με ειδικές ε, επιστηστικές ανάγκες ίσως ε, δεν ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και τα επιστημονικά πορίσματα. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μια απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων. Αξιέπαινο αυτό. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και να διαμορφώσουμε καλύτερα και πιο αυστηρά τις νομοθετικές διατάξεις μας, να απαγορεύσουμε την, την παρουσία φυτοφαρμάκων σε τροφές που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ή για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Είναι αρκετά περίπλοκη η νομοθετική ρύθμιση που έχουμε στον τομέα αυτό. Οπότε απομένει το ερώτημα και πάλι τι θα συμβεί με τροφές για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκι και τι θα συμβεί με το υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος, το ε, γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας. Δεν προκύπτει με σαφήνεια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως τα επιστημονικά πορίσματα και, και την επιρροή που έχει η παρουσία φυτοφαρμάκων σε, στον ανθρώπινο οργανισμό και ανάλογα να, λάβουμε κάποια μέτρα. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αντελάνη για την εργασία που έκανε εν ονόμα της πολιτικής μας ομάδος αλλά πέραν της σημασίας της συζητήσεως για τις ε, βρεφικές τροφές υπάρχουν και άλλα θέματα σημαντικά διότι 10 έως 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από δυσανεξία λακτόζης ή φρουτόζης και η σταμίνης και πιστεύω ότι οι, οι ιατροί είναι της γνώμης ότι η αριθμή αυτή είναι πολύ πιο υψηλή. Άρα καταρχήν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και για τους ελεγκτές αλλά και για τις εταιρείες που παράγουν τέτοια προϊόντα και για τους καταναλωτές να καταλάβουν τι αγοράζουν διότι τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει πάρα πολύ και υπάρχουν πολλά προσθετικά ε, διατροφικά ε, με βιταμίνη C παραδείγματος χάρη για ε, ηλικιωμένους ή για άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος πάρα πολύ γρήγορα και προσφέρονται διάφορες λύσεις. Όλα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται διότι η νομοθεσία σχετικά με τα βρεφικά γάλατα, τα τρόφιμα για ειδικούς, ε, ειδικές κατηγορίες ε, ασθενών. Πόσο θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σαφή σήμανση και ότι θα μπορούμε ε, και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και πώς θα μπορούν οι αρχές να ελέγχουν διότι πρέπει να δούμε δυστυχώς ότι όταν όλα αυτά μετατραπούν σε εθνική νομοθεσία δεν γίνονται σεβαστές οι αρχές αυτές. Ευχαριστώ. Η κυρία Westling. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτω με ό,τι είπαν πολλοί εκ των προληψάντων συναδέλφων. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε ε, από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην αγορά του πιο ευάλωτους ε, καταναλωτές. Ε, Βεβαίω θα πρέπει να προστατευτούν και αυτοί που έχουν δυσανεξία στην γλουτένη. Ξέρετε είναι καλύτερα να συμπεριληφθούν και τα προϊόντα αυτά ή κάποια προϊόντα γενικά στον κανονισμό παρά να αναγκάσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Ε, πιστεύω ότι ε, ε, έχουμε αυτό το πρόβλημα του, της τροπολογίας 86. Η Έστερ Ντελάγκε θεωρεί ότι πρέπει να έχει κανείς παιδιά για να έχει άποψη. Εγώ έχω δύο παιδιά βέβαια τα οποία εθήλασα αλλά παρόλα αυτά ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τα γάλατα των διαφόρων ε, κατηγοριών ηλικίας. Ε, ε, αλλά ξέρετε, είναι, πολύ είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτεί κανείς διαβάζοντας τα κουτιά με τα γάλατα για πρώτη, δεύτερη βρεφική ηλικία. Είναι τόσο περίεργες οι ενδείξεις που δίνονται που μπορεί να, να υπάρξει εύκολα σύγχυση. Και να σας πω ότι και εγώ μερικές φορές παρά τις γνώσεις μου έχω αγοράσει πράγματα κατά λάθο. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό η κυρία Κλάσσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα τρόφιμα, δηλαδή το μέσον για επιβίαση, είναι πολύ σημαντικό και μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως τα τρόφιμα για τα βρέφη, διότι θα βοηθήσουν και στην ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν κίνδυνοι επ' αυτού, διότι πολλοί κατασκευαστές έχουν συνδυάσει το όνομά τους με τα προϊόντα αλλά κάθε έξαρση θα πρέπει να τιμωρείται διότι έχουμε για τα φυτοφάρμακα αυστηρή νομοθεσία που ισχύει από πέρυσι και ιδίω όσον αφορά ε, τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων είμαστε σε πολύ χαμηλότερες τιμές αλλά κανένας έλεγχος δεν μπορεί να αποδείξει αν κάποιο φυτό έχει επηρεαστεί από φυτοφάρμακα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους. Υπάρχουν όμως αδύναμες και βάλλοντες ομάδες όπως ε, τα ε, βρέφη και οι ηλικιωμένοι οι οποίοι χρήζουν βοηθείας, η οποία πρέπει να βελτιωθεί και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αναλάβουμε στις ευθύνες μας και στην Ολομέλεια ευχαριστώ την εισηγήτρια και την δικιά μας σκιώδη εισηγήτρια την Έστερ Ντελάνια για την εξαιρετική εργασία. Αλλά θα πρέπει τα παιδιά άπαξ και γίνουν ενός έτους να μπορούν να τρώνε στο τραπέζι με την οικογένεια και να μεγαλώνουν κανονικά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Σπυρίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια ε, και τους σκιώδη εισηγητές ε, για τις ε, συμβιβασμούς τους οποίους επέτυχαν στην ΕΜΒ. Αυτό σημαίνει ότι θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε μεγαλύτερες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών. Ε, στην αρχική πρόταση δεν μπαίνουν τα προϊόντα χωρίς γλουτένη και αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται πρόβλημα για μια κατηγορία ανθρώπων, ανθρώπων ε, που έχουν πρόβλημα με την ε, ουσία αυτή και επομένως θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά την διατροφή τους στην, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μπορούμε να προτείνουμε ε, μία οριζόντια διευθέτηση βάσει του 1169 του 2011 ε, και όσον αφορά ε, προϊόντα χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες και βεβαίως έτσι ώστε μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού να έχουν την σωστή διατροφή. Για ένα λεπτό το λόγο κυρία Κάντενμπαχ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι ε, η ρύθμιση την οποία εξετάζουμε επιτυγχάνει τους στόχους που επιζητούμε, δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια για τους παραγωγούς, για τους ε, καταναλωτές και καλύτερη δυνατότητα ελέγχου. Ήδη γίνεται ένα βήμα για την ε, βελτίωση της δυνατότητας επιλογής στον χώρο των τροφίμων, αλλά υπάρχουν διάφοροι καταναλωτές καταναλωτές οι οποίοι πρέπει να καλύψουν στην αγορά και τις ιατρικές τους ανάγκες. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες, ιδίως εάν πρόκειται ε, για ασθενείς καρκινοπαθήσεις ή με άλλες σοβαρές παθήσεις. Χρειάζεται όμως και ασφάλεια για τα βρέφη, για τους, τις νεότερη γενιά και θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, τι δεν, δεν ενδείκτηται να καταναλωθεί καταναλώνεται από τα βρέφη και ε, που εριλαμβάνεται στις βρεφικές τροφές. Αυτό όμως ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, αλλά δεν μπορεί να καλύψει και προϊόντα τα οποία δεν απευθύνονται σε αυτή την ηλικία. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ είμαι υπέρ της έκθεση κυρίας Σερή για την πρόταση κανονισμού που θα αναθεωρήσει και θα συμπληρώσει τους κανόνες για τα τρόφιμα που προορίζονται σε βρέφη, μικρά παιδιά και για ειδικού ιατρικούς σκοπούς. Γιατί θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πιο σαφές και συνεπές νομικό πλαίσιο να δώσουμε έμφαση στην υποχρέωση χορήγηση ε, τεκμηριωμένων και αντικειμενικών πληροφοριών ε, προ καταναλωτέ. Και έχουμε το θέμα τη διαφήμιση για τα βρεφικέ τροφέ μέχρι 6 μήνε ε, και για παιδιά μέχρι 2 έτη. Γιατί πολλέ φορέ οι παραπλανητικέ διαφημίσει μπερδεύουν του γονεί και τους κάνουν θύματα του μάρκετινγκ αντί να έχουν στη διάθεσή τους επιστημονικά πορίσματα και σαφείς γνώσεις για να έχουν σαφή γνώση και να αποφύγουν οποιοδήποτε κίνδυνο στην επιλογή των τροφίμων. Τέτοιος κίνδυνος θα πρέπει να αποσοβηθεί με αυστηρότερους ελέγχους. Πιστεύω ότι η έκθεση θα μπορούσε να προβλέψει και μηχανισμούς ε, πιο αποτελεσματικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να γίνεται εκ των προέρων ε, αλλά με βάση μια συνολική αξιολόγηση που θα γίνεται με, όλα τα συστατικά, με βάση όλα τα συστατικά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την συγκεκριά μας για την ε, εξαιρετική έκθεση που υπέβαλε. Ε, ήρθε επιτέλους η ώρα να βελτιώσουμε την ομοθεσία για τέτοιες ειδικέ τροφέ, γιατί πολλές φορές ε, η επιστηστική βιομηχανία αναπτύσσεται πολύ πιο ραγδαία από την νομοθεσία που την παρακολουθεί. Πολλοί ε, άνθρωποι πάσχουν από όλο και περισσότερες ασθένειες θα πρέπει λοιπόν να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουμε υπόψη ε, τις ειδικέ ανάγκες πιο ευάλωτων ανθρώπων όπως είναι οι αλλεργικοί ή οι πάσχοντες από διάφορες ασθένειες. Δεν είναι πολύ εύκολη η ε, ε άντληση κάποιων πληροφοριών. Για το γάλα δεύτερη ε, βρεφική ηλικία βλέπουμε μεγάλα γράμματα 1, 2, 3, αλλά πολλέ φορέ οι γονεί αγοράζουν σπιωσμένα. Και εμένα μου έτυχε και χάνονται μέσα σε αυτή την πληθώρα πληροφοριών και διαφημιστικών πληροφοριών που λαμβάνουν. Θα πρέπει στη συσκευασία να παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο οι πληροφορίες, να δίνονται σαφείς πληροφορίες προς τους γονείς για να ξέρουν τι ακριβώς αγοράζουν οι γονείς. Αυτό δεν έχει σχέση με τη διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι σημαντική. Αλλά και για τη διαφήμιση θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, γιατί πολύ συχνά οι ισχυρισμοί υγείας είναι εσφαλμένοι ανεδαφική. Αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση στους καταναλωτές. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της νανοτεχνολογίας. Ε, οι νανοτεχνολογίες και τα νανοηλικά έχουν όλο και μεγαλύτερη παρουσία στην παρασκευή τροφών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στις νανοτεχνολογίες προκειμένου να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους ε, συμπολίτε μα. Ευχαριστώ. Στο Κάτσι τώρα, η κυρία Ράις Γκέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο μέσος καταναλωτής μπορεί ε, να καταναλώνει όλα τα προϊόντα που περιέχει ε, ένα ε, κατάστημα τροφίμων αλλά για οι ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών χρειαζόμαστε ιδιαίτερες διατάξεις για τη σήμανση των τροφίμων. Έχοντας και εγώ παιδιά πιστεύω ότι δεν πρέπει να ομορφωθούμε φαίνουμε την συσκευασία των τροφίμων κατά τρόπον ώστε να νομίζει κανείς ότι είναι καλύτερα από την πραγματικότητα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ το γάλα που προαναφέρθηκε γιατί γλυκίζει και δεν είναι η σωστή γεύση στην οποία πρέπει να εθιστούν τα παιδιά. Για τη γλουτένη χρειαζόμαστε σοβαρή, ε, σοβαρή ε, παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από αυτήν την ε, δυσανεξία και καλό ήταν ότι περιλάβαμε τη δυσανεξία αυτή στον κανονισμό κατά τρόπον ώστε ε, να μπορούν τα άτομα αυτά να αντικαθιστούν την έλλειψη της γλουτένης με διάφορες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τη Φρεντερή Κρίς για την αξιέπαινη προσπάθειά της και την εξαιρετική έκθεσή της. Ήταν επιτέλους καιρός να ρίξουμε λίγο φως σε μια κατάσταση που ήταν αρκετά συγκεχημένη για να προστατεύσουμε τις ευπαθέστερες ομάδες του πληθυσμού. Ε, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην επιστηστική βιομηχανία αλλά να μην ξεχνούμε και τη δημόσια υγεία. Δεν διεκδικούν κάποιες αλλαγές ε, στη σήμανση. Στο παρελθόν ε, ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνει κανείς επιλογή. Ήξερε τι είναι καλό και τι όχι για τα παιδιά. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν δίνεται πληρο... περισσότερες πληροφορίες στο θέμα της διαπαιδαγώγησης. Ε, γιατί πολλές φορές τα παιδιά είναι ο στόχος της διαφήμισης και πολλές φορές τα παιδιά δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα προϊόντα, πώς παρασκευάζονται, ποια είναι η προέλευσή τους. Καλό θα είναι να δοθεί έφαση όχι μόνο στις εμπορικές δραστηριότητες αλλά και στις, ε, στη διαπαιδαγώγηση για να ξέρουν τα παιδιά τι καταναλώνουν. Μια καλή διαπαιδαγώγηση, μια καλή πληροφόρηση και ενημέρωση θα αποβεί προς όφελος όλων τελικά. Πότε επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες για καλύτερη ενημέρωση και των νέων και των παιδιών για να διαμορφώσουμε μια, έναν όλο και υγιέστερο ευρωπαϊκό πληθυσμό με σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφόσον ε, το ε, ε, στομάχι μπορεί να αφομοιώσει τα τρόφιμα μόνο μετά από δύο-τρεις μήνες θα πρέπει η διατροφή των βρεφών να χρήσει ιδιαίτερη προσοχής και το λέω γιατί έχω πέντε παιδιά. Έχουμε διάφορες απόψεις σχετικά με διάφορα θέματα θέματα και ε, πιστεύω ότι ε, δεν ε, συμφωνούν όλοι για το πόσο πρέπει κανείς να τρέφει τα βρέφη. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει ο κάθε γονιός να αποφασίζει μόνος του τι είναι σωστό για τα παιδιά του και αυτό είναι προφανές θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει όλα τα, όλες τις διαφημίσεις οι οποίες θα αποκλίνουν τους γονείς από το στόχο αυτό αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Κάλενμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, εδώ θα ήθελα να προσθέσω και μία παράκληση διότι συζητάμε και το πολιετές πρόγραμμα ε, υγείας και ε, εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς και θα πρέπει να συνδυάσουμε το θέμα της παιδείας. Θα πρέπει όλοι να μπορούν να διαβάζουν τις σημάνσεις αυτές διότι δεν υπάρχει νόημα κάποιος να μην γνωρίζει ε, τι αγοράζει αν δεν γνωρίζει τι είναι οι προσωπικές του ανάγκες και γι' αυτό πιστεύω ότι στο σημείο αυτό χρειάζεται να μπορεί να υπάρχει η αναγκαία παιδεία σχετικά με την υγεία η οποία να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Κύριο κύριος Σλίτερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι θεωρούμε ότι υπάρχει μια απλούστευση ε, ε, όσον αφορά αυτές τις ε, κατηγορίες γάλακτος, αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ηλικιακή όσον αφορά αυτό το, το γάλα. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και τελικά αυτό το γάλα τι είναι. Είναι αγελαδινό γάλα στο οποίο έχουν προσθεθεί κάποια άλλα στοιχεία έτσι ώστε να καλυφθεί καλυφθούν κάποιες ε, ειδικέ ε, ανάγκες. Έχουμε επίσης και κάποια άλλα ε, τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά γευμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά ειδικά τρόφιμα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Δάλη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι οι απόψεις μας ε, προσωμιάζουν όσον αφορά την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων μερίδων του πληθυσμού. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά που ακούστηκαν στη συζήτηση αυτή όσον αφορά το ζήτημα των ειδικών κανόνων για τα γάλατα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν διεστάμενες απόψεις σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Παρ' όλα αυτά ε, θα πρέπει να ζητήσουμε την, ε, μια γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ όσον αφορά ε, τα γάλατα αυτά θα φροντίσω να γίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει βεβαίως να δούμε και το θέμα της παραπλανητικής διαφήμισης ή της ειδική διαφήμισης όπως ανέφερε το θέμα αυτό η κυρία Βίτλοκ. Όσον αφορά το ζήτημα των φυτοφαρμάκων, συζητήθηκε αυτό το θέμα πρόσφατα και λαμβάνει υπόψη τις ευάλωτες ομάδες, ειδικά δεν τα παιδιά. Ε, συμφωνώ ότι τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να περιοριστούν στη χρήση τους ε, όσον αφορά ε, προϊόντα τα οποία τελικά θα καταναλωθούν από βρέφη και μικρά παιδιά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ήδη για τις βρεφικές τροφές και τις παιδικές τροφές προβλέπονται πολύ χαμηλά αν όχι μηδενικά ποσοστά φυτοφαρμάκων. Πρέπει όμως εδώ να σας πω το εξής. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε την εφαρμογή και την παρουσία των φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει να περιοριστούμε στην απαγόρευση της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε την παρουσία φυτοφαρμάκων ε, ε, χωρίς όμως να ε, καλύπτουμε την, το ενδεχόμενο ήδη προσβεβλημένων αγρών που μπορεί να οδηγήσουν σε παρουσία φυτοφαρμάκων ε, στις ε, ε, τροφές. Αυτό που θα πρέπει να ζητήσουμε είναι η απαγόρευση της παρουσίας φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και όχι την εφαρμογή φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια. Διότι σας λέγω ότι υπάρχει ο κίνδυνος των μολυσμένων αγροτεμαχίων. όσον αφορά ε, την εντύπωση ότι η πρότασή μας προσπαθεί να μειώσει ε, την ε, προστασία ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκά. Και από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να αυξήσουμε αντιθέτως την προστασία των ανθρώπων αυτών διατηρώντας τους κανόνες όσον αφορά την αναφορά των συστατικών και την σύσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση και και μάλιστα θέλει να μεταφέρει όλα τα στοιχεία αυτά σε μια άλλη οδηγία η οποία αφορά την πληροφόρηση ε, για τα ε, προϊόντα διατροφής ε, έτσι ώστε να προστατεύσει ανθρώπους που πάσχουν από την ασθένεια αυτή. καλύτερα προστατεύονται εάν δεν αναφερθούν στην συγκεκριμένη οδηγία αλλά στην οδηγία για την πληροφόρηση ε, για, τον, ε, ε, για την πληροφόρηση των τροφίμων. Επίσης, ε, τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται σε ανθρώπους με δυσανεξία στην ε, γλουτένη ε, και αυτά καλύπτονται καλύτερα στην οδηγία για την σωστή πληροφόρηση όσον αφορά τα προϊόντα διατροφής. Καλύπτονται καλύτερα εκεί, γιατί εκεί λέμε ότι θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η περιεκτικότητα ή το ενδεχόμενο περιεκτικότητα σε γλουτένη. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία για δυο λεπτα η κυρια ριση σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες συμπερασματικές ε, παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, πήραν τον λόγο γιατί σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι διεφάνει μια συνολική ε, στήριξη της ε, ε, συμβαστικής πρότασης πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια μεγάλη ποικιλία παρεμβάσεων μπορούν να υπάρχουν και διαφορετικές αποχρώσεις όσον αφορά την σήμανση και την ε, ε, τη διαφήμιση. Βεβαίως ε, είναι πολύ σωστά αυτά που είπαν οι ομιλητές όσον αφορά τα γάλατα πρώτης δεύτερης βρεφικής ηλικίας και η κυρία Ντελάνγκη αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Λούιτερ είναι και δικό, δικιά μου ανησυχία. Η, το θέμα της ύπαρξης φυτοφαρμάκων, παρουσίας φυτοφαρμάκων βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε σε πιο φιλόδοξους στόχους, σε πιο εξειδικευμένους στόχους που θα αφορούν ακριβώς εξειδικευμένες ομάδες πληθυσμού. Και φυσικά το κείμενο θα πρέπει να είναι συνεκτικό και με την, και με την κάθετη και εγκάρσια νομοθεσία. Ε, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε πρώτη ε, ανάγνωση. Κρίμα που η Προεδρία δεν εκπροσωπείται εδώ, γιατί είναι εν μέρη και δικό της ε, ε, σφάλμα και πάντως φαίνεται ότι εδώ διαφέρονται και τα όρια της διαδικασίας που έχουμε ακολουθήσει από το 2009 όπου το Κοινοβούλιο και οι φιλοδεξίες του Κοινοβουλίου δεν ε, ανταποκρίνονται πάντα ή μάλλον δεν καλύπτονται πάντα από την διαδικασία αυτή. Ελπίζω ότι η δεύτερη ανάγνωση θα είναι γρήγορη και θα ακολουθήσει τη σωστή ορθή ε, διαδικασία. Ε, έχουμε δύο σημεία ε, που μας διαφοροποιούν από την Επιτροπή. Πρώτον, τα προϊόντα χωρίς ε, γλουτένη ή ε, παραπομπή στην νομοθεσία Food Information, πληροφόρηση για, για τα τρόφιμα, δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετή όσον αφορά την ασφάλεια και την εγγύηση των, της σύνθεσης. Αλλά βεβαίως και αναφέρατε στην αρχή της παρέμβασής σας της κατεξουσιοδότησης πράξης εμείς Οπωσδήποτε σαν κοινοβούλιο θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, θα ασκήσουμε το δικαίωμα εποπτείας το οποίο έχουμε. Πρόκειται για θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά ε, και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν γρήγορα και υπό ε, Κυπριακής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ρης. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 12. Παίρναμε στο επόμενο θέμα. Δηλαδή τα αποθέματα Ρέγκας στα δυτικά της Σκοτίας. Και μια και πρόκειται για Σκοτία, αρμόδιος συγητής είναι ο κύριος